Το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης είναι οι διαβουλεύσεις για την αναστολή της συμφωνίας της Κοτονού στην προς την Ουγκάντα και την Νιγηρία μετά την πρόσφατη νομοθεσία που κολλάζει με πολύ αυστηρό τρόπο την ομοφιλοφιλία. Θέλω να <clears throat> πληροφορήσω τους συναδέλφους ότι από μεθαύριο στο κτίριο αυτό θα συνεδριάσει η ισομερή συνέλευση των χωρών και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μια συνάντηση που κάναμε σήμερα το πρωί τα μέλη από την ευρωπαϊκή πλευρά του Προεδρείου της Ισομερούς Συνέλευσης αποφασίσαμε ότι το κείμενο το οποίο θα εγκριθεί στην σημερινή συζήτηση θα είναι και το σημείο αναφορά της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που θα αντιμετωπιστεί στην ε, ισόμερη συνέλευση, όπου φυσικά είναι παρούσες και η Ουγγάντα και η Νιγηρία. Έχει το λόγο του ο συντάκτης του ψηφίσματος, όπως άλλοι πέντε συνάδελφοι, ο κύριος Τάνοκ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ο πρόεδρος της Ουγγάντα, Γιαβέρη Μουζαβένη, πήρε απόφαση πρόσφατα να εφαρμόσει πολύ σκληρά, σκληρή νομοθεσία κατά των ομοφυλοφίλων και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό. Μεταξύ από τις λαμπρές του ρήτρε είναι φυλάκιση διαβίου για το έγκλημα της άγριας ε, ομοφυλοφιλίας μαζί με την ε, έγιναν και πιο αυστηροί οι νόμοι στην Ιγυρία από τον πρόεδρο Τζόναθαν. Οπότε τελικά είναι απογοητευτική αυτή η διάκριση που βλέπουμε κατά απλών ανθρώπων που μόνο σε έγκλημα είναι ότι ελκύονται από κάποιον του ιδίου φίλου με αυτού. Απορρίπτουν την κατηγορία του κατά κάποιο τρόπο. Είναι εισαγωγή από, την, από τι απικίε. Ε, είναι ευαίσθητο θέμα και πρέπει να προσέξουμε στην απάντησή μας να μην αποξενώσουμε τις κυβερνήσεις και να μην αποτρέψουμε το διάλογο, αλλά να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αναστολή τη Συμφωνία του Κοτονού και η βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ενώση μπορεί να πηγαίνει πιο πολύ προ μη κυβερνητικέ οργανώσει παρά προ κυβερνήσει. Αυτό πάντα το έχουμε στο πρόγραμμά μα, διότι εμεί πρέπει να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλου ανεξαρτήτω φύλου. Ευχαριστώ πολύ. Ο συντάκτη, ο κύριο Ραούλ Ρωμέβα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Για μια ακόμη φορά πρέπει να καταδικάσουμε των ε, τις, ε, τους νόμους ε, στην Ιγυρία και στην Ουγκάντα που παραβιάζουν το δικαίωμα έκφρασης, συνέρχεστε, συνεταιρίζεστε και την προστασία από απάνθρωπη μεταχείριση. Τα θέματα του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας του φύλου είναι ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη δυτική σφαίρα και τα εγγυώνται οι διεθνείς συμβάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων ε, ΛΟΑΔ. Η Νιγηρία και η Ουγγάντα δεν πληρούν με τους νόμους αυτούς ε, το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και το κράτος δικαίου. Και αυτά τα αναφέρει το άρθρο 2 της Συμφωνίας Κοτονού, πρέπει να τηρούνται αυτά τα... Ε, γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ξεκινήσουν δυνάμει του άρθρου 96 της Σύμβασης Κοτονού, να ξεκινήσουν λοιπόν διαβουλεύσεις με τις δύο αυτές χώρες με στόχο την αναστολή ε, της συμφωνίας, εάν δεν άρουν αυτά, αυτές τις αποφάσεις. Πρόεδρος, για δύο λεπτά ο συντάκτης έχει τώρα το λόγο ο Ζαρέπο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό είναι ένα ψήφισμα ε, για το, με το οποίο ζητάμε να γίνεται σεβαστή η Οικουμενική Αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιόνται ίση. Κανείς δεν μπορεί να ζει στο φόβο λόγω της σεξουαλικής του προτίμησης. Παρά το γεγονός αυτό όμως, ακόμη και σήμερα σε 76 χώρες θεωρείται έγκλημα η ομοφιλοφιλία. Σε 5 δε ε, από αυτές τις χώρες μπορεί κανείς να καταδικαστεί σε θάνατο. είναι ε, απαράδεκτες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ε, οι αποφάσεις της Ουγκάντας και της Νιγηρίας και παραβιάζουν και την συμφωνία του Κοτονού με την οποία ενώ Ένωση παρέχει ένα πλαίσιο στις χώρες ΑΚΕ για να αναπτύξουν την κοινωνία, την οικονομία τους, ε, τον πολιτισμό τους. Για καλό λόγο Ζητούμε από την Κομισιόν ε, να ξεκινήσει αυτές τις πολιτικές διαβουλεύσεις για αναστολή της Συμφωνίας του Κοτονού, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία. Πρέπει την αναπτυξική βοήθεια να ε, την στρέψουν σε διαφορετική κατεύθυνση, όχι στις κυβερνήσεις των δύο χωρών, αλλά σε ΣΜΚΙΟ. Και αυτή τους απόφαση είναι θετική. Βέβαια, δεν θέλουμε να ανασταλεί η βοήθεια, αλλά να δοθεί πιο αποτελεσματικά, να αλλάξει κατεύθυνση. Πρέπει να προστατεύσουμε τους ε, ανθρώπους ΛΟΑΔΜΕ και πρέπει να δράσουμε με βάση τις δεσμεύσεις μας. Θα πρέπει ε, να βγει από το ποινικό δίκαιο η ομοφιλοφιλία. Στην ε, και στην Ουγκάντα. Η Νιγηριανοί αλλά και άλλο δαπεί στην Νιγηρία κινδυνεύουν να συλληφθούν αν είναι ε, νομοφιλόφιλοι ή ακόμη και να δεχθούν ε, επιθέσεις. Πρέπει να τηρήσουν λοιπόν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις αυτές οι δύο χώρες. Πρόεδρος, ο συντάκτρο ψηφίσματος για 1,5 λεπτό τώρα έχει το λόγο κυρία Σάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσει εδώ την Κυριακή η συνέντευξη εκπροσώπηση ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει ε, οι νόμοι τη Νιγηρία και τη Ουγγάντα για την ποινικοποίηση τη ομοφιλοφιλία να ε, συζητηθεί. Γιατί είναι αυστηρέ οι ποινέ που επιβάλλονται, παραβιάζεται η συμφωνία του Κοτονού και έχουμε ε, το άρθρο 96, την ανθρωπιστική ρήτρα, ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να αντιμετώπισουμε αυτό το θέμα. ποινικοποιούνται οι με μια εμπνεόμενη από την άκρα συντηρητική αμερικανική ε, υπερθρησκευτική ιδεολογία. Τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να, κάποια από αυτά να παγώσουν την αναπτυξική τους βοήθεια κάτι μεν ανεπιθύμητο αλλά αναγκαίο όπως κρίνουν. Επιθυμία μας δεν είναι βέβαια οι απλοί άνθρωποι να υποφέρουν περισσότερο από ό,τι ήδη υποφέρουν σε αυτές τις αφρικανικές χώρες. Τα προβλήματα όμως επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο. Είναι η διαφθορά, οι κακές υποδομές, ανάγκη μεγαλύτερης ανάπτυξης, παιδείας, η ανάγκη να πάψει ο βίος εξτρέμισμος. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε τον ενεργό μας διάλογο και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε μεν, αλλά χωρίς ε, να απεμπολίσουμε τις αρχές, τις αξίες μας και τις δεσμεύσεις μας ε, και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ε, με τις αμοιβές συμφωνίες και οι δύο αυτές χώρες. Και πρέπει να δεσμευτούν ότι θα σέβονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόνικ για ένα λεπτό και αυτός συντάκτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαστε αποφασισμένοι να δραστηριοποιηθούμε όσον αφορά την Ογκάντα και την Ιγυρία και θέλουμε να καταδικάσουμε και τους νόμους που υιοθετήθηκαν το Δεκέμβριο. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή χώρες με τις οποίες εργαζόμαστε πολιτικά και έχουμε ε, σχέσεις εμπορικές και στέλνουμε αναπτυξιακή βοήθεια να παραβιάζουν σε τέτοια κλίμακα τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως βλέπουμε να συμβαίνει στην Ουγκάντα και την Ιγυρία. Μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα την ποινή φυλάκιση δεκαετούς κάθριξης που αποφασίστηκε για εκείνους που ε, ε, συναντήθηκαν στα πλαίσια μιας οργανώσεως που εξυπηρετούσε την κοινότητα των ΛΟΑΔ. Σε 12 επαρχίες της Νιγηρίας οποιαδήποτε ομοφιλοφιλική επαφή σημαίνει ότι κάποιο άτομο μπορεί να τύχει και της ποινή, της θανατικής ποινής. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν Ευρώπη, έχουμε κυρώσει που μπορούμε να επιβάλλουμε στα πλαίσια της Συμφωνίας Κοτονού και καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει να παρέμβει κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που θα λάβει η χώρα. Ε, Τελευταία παρέμβαση από την συντάκτρια, την τελευταία συντάκτρια της κυρίας Βερζιά, που έχει δύο λεπτά για την παρέμβασή της. Η Ουγγάντα ε, υπήρχε τα προβλήματα, ο πρόεδρος Μουσεβένη τελικά στις 24 Φεβρουαρίου πέρασε το νόμο που ποινικοποιεί την ομοφιλοφιλία. Η θανατική ποινή μετάλλαξε σε ισόβια κάθυρξη. Ε, λοιπόν, δεν μπορεί να, να σκοτωθεί λοιπόν, δεν μπορεί να το σκοτώσουμε η πρόεδρος. Στην Ιγυρία επίσης έγινε το ίδιο, πέρασε ανάλογος, μήνας, ανάλογος νόμος στις 13 Ιανουαρίου και ε, μαστιγώθηκε ένας που καταδικάστηκε 15 φορές. Ήταν η δύσκολη κατάσταση, η δημοφιλοφιλία ήδη ε, κατεστέλετο βιαίως. Σήμερα περνάμε κάποιο στάδιο και πιστεύετε ότι μπορεί να διώκονται δημοφιλόφιλοι κυρίως οι καθολικές και οι αμερικανικές εκκλησίες έχουν προφανώς αρνητική επιρροή ε, στον πληθυσμό. Υπάρχει κλίμα έντασης ε, που ισχύει και διάφορες εφημερίδες, φυλάδες εντόπισαν 200 ονόματα ομοφιλοφίλων με ονόματα και φωτογραφίες. Και μια πρώτη φυλάδα που δημοσιεύθηκε το 2011 κόστισε τη ζωή στον ε, κάτω Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που τροφοδοτεί το μίσος. Είναι αόριστη η όρη της νομοθεσίας. Όλοι μπορούν να εμενεύσουν τον νόμο όπως θέλουν. Ε, πάντα όταν υπάρχει αόριστο νομικό ε, μπορεί να το εκμεταλλευτούν. Λοιπόν, θέλουμε, δεν μπορούμε να δεχόμαστε συμφωνία κοτονού χώρες που έχουν τέτοιες νομοθεσίες. Η Ουγγάντα, η Νιγηρία θα πρέπει να καταργήσουν την νομοθεσία που παραβιάζουν τις διεθνείς τους ε, υποχρεώσεις. Πρέπει να πιέσουμε τις χώρες αυτές εφαρμόζοντας το άθρο 96 της Συμφωνίας Κοτονού, υποστηρίζοντας και δημοσία πολιτικά και οικονομικά τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Θα πρέπει να γραμμίσουμε σε ποιο βαθμό η μπλοκή τους επιτόπου είναι απαραίτητη για να υπάρξει πραγματική αλλαγή νοοτροπίας και να φύγει ο σκοταδισμός από όπου και να προέρχεται. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές του Κοτονού Λοιπόν, θα πρέπει τελικά να προσπαθήσουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση. Κριστίν. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα τους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών τους ομάδων. Για δύο λεπτά ο κύριος Βον για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Νιγηρία και η Ουγγάντα Υιοθέτησαν νόμους που ποινικοποιούν όλο και περισσότερο την ομοφιλοφιλία και γύρονται και συνομιλίες, οι λόγοι και για παρόμοια προβλήματα σε άλλες χώρες. Επί σειρά ετών δημιουργείται αυτή η κατάσταση, εξελίσσεται και τώρα είναι πραγματικότητα. Πολλοί βέβαια θα υποψιάζονται ότι αυτοί οι νόμοι θεσπίζονται από πολιτικού ηγέτε που θέλουν να προσερκίσουν την προσοχή του σε άλλα προβλήματα, να τα απομακρύνουν την προσοχή από τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σιωπά επ' αυτού και θα πρέπει να δείξει ότι είμαστε σοβαροί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι η λύση θα πρέπει να προέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από μεμονωμένα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στο εγγύς μέλλον όπου θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πέρα από την εκκίνηση διαβουλεύσεων σχετικά με τη συμφωνία υπάρχει η ισομερή συνέλευση ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρατε κύριε Πρόεδρε και θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία να θέσουμε το ζήτημα εκεί. Υπάρχει και πολιτικός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει προγραμματιστεί με την Ογκάντα στις 28 Μαρτίου και υπάρχει η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ενώσης Αφρικής στις 2 και 3 Απριλίου. Υπάρχουν δυνατότητες για να θέσουμε το ζήτημα. Κάποιοι από εμά αναφερθήκαν και στην αναστολή της παροχής ε, βοήθειας σε αυτές τις χώρες. Προτιμότερο θα ήταν, όπως είπαν και άλλοι, να κατευθυνθούν περισσότερα χρήματα προ μη κυβερνητικέ οργανώσει, κυρίω προ εκείνε που ασχολούνται με παιδεία και υγεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση πιστεύω θα πρέπει να παροτρύνει την Αφρικανική Ένωση να αναλάβει το θέμα και να δείξει κάποια ηγετική προσέγγιση ούτω ώστε το ζήτημα αυτό να μην διαδοθεί και η προσέγγιση να διαδοθεί σε όλη την περιφέρεια. Διότι οι άνθρωποι που και στον κόσμο αξίζουν να έχουν ανθρώπινα δικαιώματα και να υπάρχει ισοτιμία. Από τους πράσινους για ένα λεπτό η κυρία Κορνέλσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έρχεται ένα σημείο όταν πρέπει να τονίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και να το αποδείξουμε ότι είναι μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ουγγάντα και την Ιγυρία οι κυβερνήσει και τα κοινοβούλια δυστυχώ πήραν την απόφαση να ποινικοποιήσουν την ομοφιλοφιλία και του ΛΟΑΔ. Δεν ήταν μια τυχαία απόφαση, ήταν μια απόφαση η οποία ήταν ζυγισμένη και ηθελημένη. Παρά τις διαμαρτυρίες των τοπικών και διεθνών ΜΚΟ <clears throat> της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς φορείς. Τώρα οι ΛΟΑΔ της ε, Ουγκάντας μπορεί να βρεθούν στη φυλακή για χρόνια, όπως και οι φίλοι και η οικογένειά τους που τους υποστηρίζει και εξίσου τρομερή είναι κατάσταση στην Ιγυρία. Όλα αυτά οδηγήσαν σε μια αύξηση στη βία και την διάκριση κατά τον ΛΟΑΔ μόνο ένα συμπέρασμα μπορούμε να αντλήσουμε από τη δική μας πλευρά. Η Ουγγάντα και η Νιγηρία δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει της συνθήκη της Κοτονού. <clears throat> Επομένως, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την αναστολή της συμμετοχής τους και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας και την βοήθεια που δίνεται στις κυβερνήσεις αυτών των χωρών. Εάν όχι, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Κονέλσον. Τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Ομπερμάιρ για 1,5 λεπτό, εξ ονόματος τομή μη Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν σκεφτεί κανείς ότι η ομοφιλοφιλία μπορεί να τιμωρηθεί με ισόβια δεσμά στην ε, Ουγγάντα και σε χώρες όπου η Σαρία μπορεί να τιμωρηθεί με θανατική ποινή, μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο ιστερικές είναι οι φωνές για την καταπίεση των ομοφιλοφίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντλήσει τα απαραίτητα συμπεράσματα από αυτά που έχουν γίνει στην Ουγγάντα και την Νιγηρία. Δεν πρέπει η βοήθεια η οποία δίδεται να δίδεται σε κυβερνήσεις οι οποίες εφαρμόζουν τέτοιους νόμους. Δεν πρέπει να έχουν ευνοϊκές συνθήκες στο εμπόριό τους είναι μια συμφωνία, η συμφωνία με τις χώρες του ΟΑΚΕ, να ε, σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε δυνατότητα να <clears throat> δεν έχει καμιά άλλη δυνατότητα συγγνώμη στο διπλωματικό επίπεδο αλλά θα πρέπει να αντλήσει τα απαραίτητα συμπεράσματα. Το συμπέρασμα πρέπει να είναι ότι πρέπει να αποκλειστούν από τις χώρες ΑΚΕ η Ουγγάντα και η Νιγηρία. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Στην οφθαλμοσυλληπτική διαδικασία έχουμε έξι βουλευτές που ζήτησαν να λάβουν το λόγο. Και θα σας κόψω όταν φτάνει το λεπτό. Ο κύριος Σον Κέλλη έχει ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί εδώ, γιατί αυτό που γίνεται στην Ουγγάντα και στην Ιγυρία είναι απόλυτα απαράδεκτο. Ιδίω η ποινικοποίηση ομοφιλοφιλίας και οι δρακόντιες ποινέ που εφαρμόζονται. Πρέπει <clears throat> να σκεφτούμε τη βοήθεια που δίνουμε σε αυτέ τι χώρες και να σταματήσουμε να αυτή τη βοήθεια στην κυβέρνησή τους και να τη δίνουμε μόνο στις ΜΚΟ. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον πρόεδρο της Ουγγάντας, ο οποίος λέει ότι βασίζεται η απόφασή του σε μια ε, ιατρική έκθεση που λέει ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι κοινωνική, ε, δεν είναι γενετική αλλά κοινωνική συμπεριφορά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε σε ένα πιο σύντομο χρονικό διάστημα να πετύχουμε αυτό που έχουμε πετύχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρήσουμε τι νομοθεσίες μα σε λίγα χρόνια μονάχα. Η κυρία Γέγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 16 Ιανουαρίου εγκρίναμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα το οποίο καταδικάζει την απόφαση της Ουγγάντας και της Νιγηρίας να ποινικοποιήσουν την ομοφιλοφιλία. Το... <clears throat> Οι νέοι κανόνες λένε ότι οι γάμοι μεταξύ ομοφύλων, οι παριστάμενοι σε αυτούς τους γάμους και οι οργανώσεις ΛΟΑΔ θα κολλάζονται. Όλα αυτά είναι παραβίαση της γενικής δήλωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνεται στη Συνδική του Κοτονού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ω χορηγό προ τι αναπτυσσόμενε χώρε θα πρέπει να απαιτήσει οι χώρε αυτέ να σεβαστούν τα ε, οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό καλώ την Κομισιόν να αναθεωρήσει τι αρχέ συνεργασία με την Ουγγάντα και την Ιγυρία. Όλε οι μελλοντικέ συμφωνίε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτων χωρών θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ειδική ρήτρα που θα ζητήσει το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και να μην υπάρχει μια διάκριση επί τη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού. Τελείωσε ο χρόνος σας. Η κυρία Μορβάη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ροέβα και άλλοι συντάκτες ε, της εκθεσής θα ήθελαν, θα ήθελαν να απαντήσουν στο ερώτημά μου. αυτή η σταχυολόγηση, πώς γίνεται, πώς επιλέγετε και μας αναφέρετε κάποια πράγματα. Θα σας πω εγώ μια άλλη ιστορία. Ένας Σαουδάραβας διπλωμάτης ε, στη ΣΥΠΑ ε, λέει ότι είναι ομοφιλόφιλος. Απειλείται από τη Σαουδική Αραβία ότι θα βασανιστεί, θα υποπληθεί σε απάνθρωπη μετέλεση. Ζητάει άσυλο στι ΗΠΑ και οι ΗΠΑ αρνούνται να του παραχωρήσουν άσυλο. Η Σαουδική Αραβία, ισχυρή χώρα, φίλη των ΗΠΑ, η ΗΠΑ επίση μεγάλη χώρα, ακόμα και μετά τι αποκαλύψει Νόντεν πολύ καλή φίλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πολύ ωραία και ευχάριστη ατμόσφαιρα στην ε, οικογένεια αυτή. Μήπως όμως τελικά ε, κάνουμε επιλογή. Θα τεθεί αυτή η υπόθεση κάποια στιγμή υπόψη ε, του Κοινοβουλίου ή όχι. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Κόρχολα, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε πρέπει να σκεφτούμε τις αρχές της αναπτυξιακής βοήθειας και τι πρέπει να κάνουμε όταν η αποδέκτρια χώρα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η διεθνής κοινότητα δεν συγγεί. Ε, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία θα παγώσουν την βοήθεια στην Ουγγάντα ή θα την ανακατευθύνουν Κάποιοι καλό θα ήταν να κάνουν το ίδιο και για την ε, ευρωπαϊκή βοήθεια, αλλά είναι αμφίδρομο όλα αυτά. Πρέπει να στηρίξουμε τις μικρές οργανώσεις, διότι δυσκολεύονται πολύ να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς, επειδή και τα μέλη αυτών των ΜΚΟ αντιμετωπίζουν ε, την ποινή ε, το ενδεχόμενο τη ποινή να βοηθήσουν του ομοφυλοφίλου. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι όλε οι χώρε έχουν την υποχρέωση να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν τη διακριτική μεταχείριση των πολιτών του. Πρόεδρος, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μπόρις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη Συμφωνία Κοτονού και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο επιβολή κυρώσεων. Αυτό που αποφάσισαν να κάνουν οι δύο αυτές χώρες αντιβαίνει ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα παράδειγμα διακριτικής μεταχείρισης ε, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αναστείλουμε τις πληρωμές ε, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας και να στηρίξουμε τις ΜΚΟ. Αυτό θα στείλει ένα πολύ χειρό μήνυμα σε αυτές τις χώρες γιατί δεν μπορούν να παραβιάζουν κατά αυτόν τον τρόπο συμφωνίες τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια αντίδραση από τη δική μας πλευρά θα ήταν πιστεύω αποτελεσματική. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η ανθρωπιστική βοήθεια εξαρτάται και από τι δεσμεύσει που αναλαμβάνουμε όλοι όταν υπογράφουμε μια συμφωνία. Πρέπει λοιπόν όλε οι χώρε να σκεφτούν αυτό το ενδεχόμενο αναστολή πληρωμών και να δίνουν αλλού τα χρήματα στι ΜΚΟ και στι κυβερνήσει. Πρόεδρο, τελευταία παρέμβαση στο γύρο αυτών είναι η παρέμβαση του κυρίου Σιλβέστρη που έχει στη διάρκεια οι νόμοι κατά της ομοφιλοφιλίας που θετήθηκαν από την Ιγυρία και την Ουγγάντα σίγουρα είναι αδικοί και αξιοκατάκριτοι. Πρέπει να τους καταδικάσουμε και θα πρέπει να έχουμε έντονε αντιδράσει. Όμω με δυσαρεστή που βλέπω ότι σε αυτή την ευκαιρία δεν λείπουν αυτοί που εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να εισάγουν θέματα ταυτότητα του φίλου, ε, την ε, τεχνητή αναπαραγωγή δημοφιλοφίλων, ε, ζευγαριών κλπ. Διάφορα στοιχεία. Όπω αναφέρεται στα, στα, στην έκθεση πολιτικά δικαιώματα για. λοιπόν, αυτό αφορούσε τα έμβρια. Αλλά τώρα Ακούγεται η φωνή των ΛΟΑΔ, αλλά τα διάφορα αυτά τα έμβρια ποτέ δεν έχουν κάνει ακούστη φωνή. Πότε θα συζητήσουν στο δικαίωμα, το δικαίωμα των εμβρίων σε αυτό το κοινοβούλιο που είναι μια μονότητα της οποίας η φωνή ποτέ δεν ακούγεται. Ευχαριστώ κύριε Σιλβέστης. Έχουμε κλείσει και τώρα δίνουμε το λόγο στον Επίτροπο κύριο Λεβεντόφσκι για να μπορέσει να απαντήσει εξ ονομάτων της Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό που συζητούμε σήμερα είναι απλώς η νομοθεσία αυτή στην Ουγγάντα και Νιγηρία που κολλάζει την ομοφιλοφιλία. Δεν είναι φυσικά η μόνη τέτοια περίπτωση. Διάκριση εναντίον των ΛΟΑΔΜ σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια στεναρή θέση αρχής εναντίον κάθε μορφής διάκρισης. Τον Ιούλιο του 2013 το Συμβούλιο ανέκρινε νέες κατευθυντήρες γραμμές για να εξασφαλίσει τα πλήρη δικαιώματα των ΛΟΑΔ. <clears throat> Αυτό σημαίνει ίση προστασία των ομοφιλοφίλων κατά της ε, διάκρισης. Αντιμετωπίζοντας την νέα νομοθεσία στην Ουγγάντα και στην Ιγυρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει προσφυλωμένη στην αρχή της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, οποιαδήποτε πολιτιστική ή θρησκευτική ή πολιτική αξία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Και σήμερα ακόμα κάποια μέλη του Κοινοβουλίου ζητούν να εφαρμοστεί το άρθρο 96 για διαβουλεύσεις με την Ιγυρία και την Ουγγάντα. Για μας μια άμεση προσφυγή στο άρθρο 96 θα ήταν πρόορη. Έχουμε και άλλες ευκαιρίες διαλόγου και είμαστε σε πολύ ειλικρινή συζήτηση με τις αρχές και των δύο χωρών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συναντήσει τους ε, υπευθύνους της ε, Ουγκάντας και της Νιγηρίας <clears throat> για, έντονο, ενισχυμένο διάλογο στις 8 του Μαΐου. Έχουμε λοιπόν και άλλες ευκαιρίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν από τον Derek Vaughan και πρέπει να σας πω ότι από τον προϋπολογισμό μας δεν θα γίνει καμία εκταμείευση πληρωμών προς τις χώρες αυτές. Σε πρακτικούς όρους υπάρχει ένα πάγωμα των πληρωμών. Περιμένουμε από αυτές τις συναντήσεις ότι θα βγουν σημαντικά στοιχεία που θα καθορίσουν πώς οι σχέσεις μας με τις δύο αυτές χώρες, την Ιγυρία και την Ουγάντα, Ουγάντα θα συνεχιστούν επί τη βάση της Συμφωνίας Κοτονού τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι λοιπόν για να καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Έχουμε έξι ψηφίσματα για, τα, για τη λήξη της συζήτησης. Κλείνουμε λοιπόν τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει σε λίγο <clears throat> όταν τελειώσουμε και το τρίτο σημείο το οποίο θα εξετάσουμε τώρα που, που έχει να κάνει με την ασφάλεια και την ε, λαθρεμπορία ανθρωπίνων όντων στο